ξεκινήσουμε φίλοι μας, αν και είμαστε λίγοι, αλλά συνήθως είναι δύσκολο τα μέλη να καταφτάνουν στεριάτικα. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιους συναδέλφους, κάποιοι άλλοι ακόμα ταξιδεύουν. Να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη και την έγκριση της. Μία αλλαγή έχουμε. Η ψηφοφορία στο 14 για τις κοινέ διατάξεις, για τα ε, περιφερειακά ταμεία, τα ταμεία ανάπτυξης, ταμεία συνοχής και τα ταμεία ε, αλληλιάς και το καθεξής. Αυτό το σημείο τέλο πάντων το 14 αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου. Να πάμε στο σημείο 2 της ημερησίας διάταξης Ανακοινώσεις έχουμε σήμερα διερμηνία. 16 γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, δανικά. Ελληνικά μπορείτε να ακούτε και να μιλάτε στην ε, καμπίνα υπαριθμών 7 είμαστε και άλλες γλώσσες. Romania. Ε, Επίσης, έχουμε και μία ομάδα επισκεπτών στην αίθουσα, αν δεν κάνω λάθος, ή μπορεί να καταφθάνουν ακόμα. Μία ομάδα νέων από 7 ευρωπαϊκές χώρες με το πρόγραμμα Erasmus Plus και επικεντρώνεται σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Θα έχουμε και διάφορους άλλους μαζί μας στην πορεία. Α, συγγνώμη, λάθος κάνω, λέει ο Πρόεδρος. Αύριο θα καταφτάσουν. Η Αντιπρόεδρος ε, κυρία Γκέπχαρτ επίσης θα έχει προσκεκλημένους στις 20 Νοεμβρίου το απόγευμα, αύριο το απόγευμα, στο σημείο 3 της ημερής διαταξής έκθεση για τις ε, διαδεσμικές διαπραγματεύσεις, τρίτος τριμερής διάλογος για την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου στις 6 Νοεμβρίου. Και ο τέταρτος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα σήμερα το απόγευμα. Στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 9ης Οκτωβρίου. Ο κ. Μαρτάν, ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να κοιτάτε και ζητήσετε το λόγο, γιατί ξεκινήσατε ε, και είπατε ότι είναι δύσκολο να είναι εδώ πέρα οι βουλευτέ δευτεριάτικα. Είναι δύσκολο, Πρόεδρε, για ένα βουλευτή να μην καταλαβαίνει του κανόνε ή συνεδριάσει ε, τη Επιτροπή Απασχόληση ε, αναβάλλονται πλέον και καταργούνται στις Βρυξέλλες και δεν ξέρω γιατί λαμβάνουν χώρα στο Στρασβούργο. Αυτό δεν τηρεί τις ε, ιδρυτικές συνθήκες. Οι επιτροπές συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες και η Ολομέλεια συνεδριάζει στο Στρασβούργο. Και νομίζω ότι έτσι συγχαίρεται το έργο που γίνεται στο Στρασβούργο με αυτό που γίνεται στις Βρυξέλλες. Δεν μπορεί, μπορείτε λοιπόν να δικαιολογείτε τους βουλευτές που απουσιάζουν από το Στρασβούργο ή από τις Βρυξέλλες. Δεν μπορείτε να κάνετε διακρίσεις στο σημείο 1, 2 και 3. Ε, επίσης χρησιμοποιήσατε το σφυράκι σας σε ό,τι αφορά την έγκριση των πρακτικών δεν ζητήσατε ψηφοφορία. Και είναι πολύ περίεργο ο τρόπος αυτός ε, προεδρία σε μια επιτροπή. Είτε πρόκειται στι Βρυξέλλε, είτε πρόκειται στο Στρασβούργο, είτε πρόκειται για αναβολή και ε, εκ νέου ε, οργάνωση της συνεδρίαση. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί, κυρία Πρόεδρε, γιατί προφανώ στο εκλογικό μα κοινό παρακολουθεί το έργο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και τώρα μπορείτε να περάσετε στο σημείο 4 της ημερήσιας δράξης σας. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Μαρτάν. Τα σημειώνω. Τα σημειώνω όλα αυτά. Και περνάμε στο σημείο 4. Η ίδρυση του προγράμματο για την Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Ο αρμόδιο συνάδελφο ο κ. Μπονιφάη, δεν μπόρεσε να καταφτάσει εγκαίρω στις Βρυξέλλες σήμερα για την εξέταση των τροπολογιών και μου ζήτησε να πω δύο λόγια εξ ονοματός του. Οι πιο πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους στην έκθεση του κυρίας Κλούνε αποτελούν βελτίωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προθυμία για την διαμόρφωση ενός στεναρού προγράμματος για την πρόγραμμα 2020-2027 είναι σαφής και η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών υποστηρίζει πλήρως τον στόχο ενός φιλόδοξου καλοσχεδιασμένου κειμένου για το επόμενο πουδουπού. Το Ευρωπαϊκό Σώμα λοιπόν Αλληλεγγύης θέλουμε να στεφτεί με επιτυχία όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα προσέλκυσης νεαρών συμμεταχόντων και παροχής υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά πιο σημαντικά είναι ότι θα πρέπει να έχει ικανότητα να παρέχει βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται. Ένα καλοσχεδιασμένο λοιπόν κανονισμό σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, του στόχου και του μηχανισμού του μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την παροχή αλληλεγγύη σε όλα τα κρατη και εκτό αυτών. Ο κύριος Μπράντι εδώ επισημαίνει ότι κατά την άποψή του η γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης που θα υποβληθεί στους συναδέλφους από την Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ενίσχυση των, ε, του σκέλους της απασχόλησης, ιδιαίτερως μέσω της εισαγωγής κάποιων θετικών εκβάσεων και αποτελεσμάτων που έχουν τύχει επεξεργασίας με το Συμβούλιο στο παρελθόν και είναι απαραίτητο να καταρτήσουμε πιο σαφείς ε, κανόν ορισμούς για τις μαθητείες, τις πρακτικές και για τις θέσεις απασχόλησης, πάντα σεβόμενοι τις αρχές και τους όρους της απασχόλησης και των σχετικών συμφωνιών, συλλογικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών. Συμπεριλαμβανομένων ε, σωστών τρόπων προσαρμογής. Πέραν τούτου, για να υπάρχει πιο σαφής διάκριση της εθελοντικής ε, εργασίας και της επαγγελματικής εργασίας θα πρέπει να υπάρχει μια σφραγίδα διαφορετική ποιότητας για, τις δύο, για τους δύο τύπους προκειμένου να είναι σαφής η συμμόρφωση των οργανώσεων που συμμετέχουν καθώς και στις αρχές του προγράμματος. Εν γέννη υπάρχει ανάγκη το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών να καταστεί όσο πιο συμπεριληπτικό γίνεται. Καταρχάς, βάζοντας το επίκεντρο της λειτουργίας της τους οργανισμούς που συμμετέχουν και στόχος μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός προγράμματος το οποίο θα το νιώθουν δικό τους οι νέοι στο πνεύμα του Erasmus Plus. Και με τον τρόπο αυτό δίνουμε και το πιο θέλετε, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουν κρατηθεί λοιπόν ε, σχετικέ τροπολογίε προ την κατεύθυνση αυτή και ω σοσιαλιστέ και δημοκράτε ελπίζουμε ότι η συγγήτρια θα τη συμπεριλάβει στι συμβαστικέ τη τροπολογίε. Τέλο, ο Μπράντο μου ζήτησε εκ νέου να ευχαριστήσουμε την συγγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει και ζητά συγγνώμη εκ νέου για την απουσία του. Προσβλέπει στη συζήτηση με την κυρία Κλούνε και με τους Κιώδες στην επόμενη συνεδρίαση των σκεωδών την Τετάρτη το απόγευμα. Μάλιστα. Okay. Now... Μάλιστα, λέει πρόεδρος. Και τώρα να σας διαβάσω και τι λέει και η συγκύτρια. Η εισαγωγή αυτή που σας διάβασα ήταν του κυρίου Μπονιφάη, που ήταν ε, σκιώδης. Αυτό δεν το είχα λάβει από πριν. Θα προσπαθήσω να το διαβάσω σωστά. Και τώρα να μιλήσω ξανά τη κυρία Κλούνε. Uh, I'd like to... Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να παρευρεθώ στη σημερινή συνεδρίαση στην Επιτροπή λόγω άλλων υποχρεώσεων και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις υποδηματικέ τροπολογίες. Όσον αφορά την πρώτη εξέταση των τροπολογιών, αρκετές από αυτές προσπαθούν να ενισχύσουν το ε, ζήτημα της απασχολησιμότητας στην ε, άσκηση και επίσης να δημιουργήσουν μια ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά την νομοθεσία. Χαιρετίζω το γεγονό ότι οι συναδέλφοι μοιράζονται την κοινή εικόνα ότι οι ε, πρακτικές δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε την αξία που έχουν οι πρακτικές ασκήσεις για τους νέους αλλά και για τις κοινότητες ανά την Ευρώπη αλλά και αλλού. Χαίρομαι ιδιαίτερο επίσης που οι τροπολογίε επικεντρώνονται ακόμα στην ε, προώθηση δυνατοτήτων ε, για τους ε, νέους, ούτω ώστε να εκφράσουν αλληλεγγύη. Εάν όλο αυτό οδηγήσει στην ανάπτυξη ε, ικανοτήτων που μπορούν να μεταφερθούν στην αγορά εργασίας, τότε αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ αισιόδοξο και αυτό δεν θα πρέπει όμως ποτέ να οδηγήσει σε αντικατάσταση ε, των ε, θέσεων εργασιών. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να παράσχει στους νέους τη δυνατότητα ε, να μπουν σε κοινότητες, να εργαστούν και να συνεισφέρουν με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ωφέλιμος για τις πόλεις και τις περιφέρειες ενώ ταυτόχρονα θα αποκτούν νέες ε, ικανότητες και θα αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους. Οι τροπολογίες κάνουν πολλές ε, ε, θετικές παρατηρήσεις όσον αφορά τους συμμετέχοντες οργανισμούς οι οποίοι θα πρέπει να προσεγγίζουν το πρόγραμμα σχετικά με το σώμα αλληλεγγύης και ταυτόχρονα τονίζουν ζητήματα όσον αφορά τα άρθρα 11 και 12. Πολλές τροπολογίες επίσης προσφέρουν διάβγεια όσον αφορά τους ορισμούς και τις δραστηριότητες δραστηριότητες των προγραμμάτων που σχετίζονται με την Επιτροπή Απασχόλησης. Και έτσι ε, η θέση της Επιτροπής γίνεται πιο ξεκάθαρη σε όλο το κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για τους νέους Ευρωπαίους πολίτες ε, και ανυπομονώ να συνεργαστώ επικοδομητικά με συναδέλφους ε, κατά τις επόμενες συναντήσεις των σκιωδών, ούτω ώστε να παρουσιάσουμε μια καλή γνωμοδότηση από πλευράς της Επιτροπής Απασχόλησης που θα μπορέσει να προσθέσει αξία στην ε, πρόταση αυτή. Αυτή λοιπόν ήταν η εισαγωγή από την εισηγήτρια η οποία δεν μπορούσε να ήταν εδώ και Διάβασα επίσης το κείμενο του Σκιώδη, του Σκιώδη ο οποίος ε, είναι από το S&D. Υπάρχει κάποιος άλλος ε, που θα ήθελε να πει κάτι. Αρχικά το λόγο στην κυρία Ζιτνάντσκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. εξέτασα τις ε, τροπολογίες ε, των ε, συναδέλφων και συνεισφέρουν πολύ στη βελτίωση του κειμένου και ταυτόχρονα προσπαθούν με ελάχιστες βελτιώσεις να συνεισφέρουν το ώστε αυτό το κείμενο να βελτιστοποιηθεί. με αυτές τις βελτιώσεις προσπαθήσαμε και εμείς με τις δικές μας τροπολογίες να συνεισφέρουμε προς αυτό. Επίσης, ως επικεντρώθηκα εγώ προσωπικά όσον αφορά ε, στο ζήτημα της ε, προστασίας των ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να, μην, να προσέξουμε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος σε τέτοια προγράμματα δεν θα πρέπει να υποστηρίζουμε την βοήθεια οργανισμών που δεν τηρούν τα πρότυπα όσον αφορά τη, τα, τα, παγκόσμια, τα, τα ευρωπαϊκά, ε, τις ευρωπαϊκές αρχές ε, και δεν, δεν τηρούν ε, κανόνες, ευρωπαϊκούς κανόνες ε, και παρόλα αυτά να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να, επικεντρωθούμε σε δραστηριότητες οι οποίες ε, ασχολούνται και με παιδιά και θα πρέπει να απασχολούν προσωπικό το οποίο είναι κατάλληλα καταρτισμένο και ταυτόχρονα να επικεντρώνονται στην προστασία των παιδιών. Θα χαρώ λοιπόν αν υπάρξει υποστήριξη από τους συναδέλφους και θα χαρώ για τη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σελίμοβιτς από την Άλντε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Υπάρχουν αρκετά τα οποία θα θέλαμε να δούμε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την τροπολογία και γι' αυτό το λόγο θα, ε, σε αυτή την γνωμοδότηση και γι' αυτό θα καταθέσουμε τροπολογίες το συγκεκριμένο πρόγραμμα εμείς στην Άλντε υποστηρίζουμε ιδιαιτέρως, όμως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν. Αρχικά η αλληλεγγύη, απασχόληση και πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και επίσης να στοχεύσει στην αντιμετώπιση κοινωνικών ε, προκλήσεων στις ε, τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι και το όλο θέμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Επίσης, ε, η συγκεκριμένη γνωμοδότηση ε, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα ε, να τονίσει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα και σε ευάλωτες ομάδες να συμμετέχουν μετανάστες, άτομα με, ανάπη, με αναπηρία, κάτοικοι εξόχως από κεντρών περιοχών. Όλοι αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, ε, σας καλούμε να έχουμε διάφορα label ε, ποιότητας ε, και εργασίες και να μην δημιουργείται επιπλέον διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις οι οποίες ιδάλλως δεν θα συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η απλότητα λοιπόν είναι ένα βασικό συστατικό για εμάς σημαντικό επίσης ε, όσον αφορά το κομμάτι της αποσχόλησης θα θέλουμε να δούμε την αναφορά σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας της πρακτικής άξισης που θα είναι άσκησης που θα είναι έμισθη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς βλέπουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ της πρακτικής άσκησης και της εργασίας. Ναι, μπορούμε να συζητήσουμε πώς γίνεται η διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των δύο, όμως οι πρακτικές ασκήσεις θα πρέπει να πληρώνονται. Επίσης θα θέλαμε να δούμε τον ορισμό των ε, δουλειών όσον αφορά ε, την προσφορά αλληλεγγύης ε, και να αναφέρεται στους τρεις μήνες και όχι στους δύο μήνες. Και τέλος θα θέλαμε και θα επιστρέψουμε σε αυτό με τροπολογίες πάνω σε αυτό το θέμα και θα χαρούμε να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες ομάδες πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπόιλαν από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν ήταν πιο ξεκαθαρό, δεν θα υπήρχε σύγχυση σχετικά με το τι συμβαίνει στι Βρυξέλλε και ε, το Στρασβούργο. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη και την πρώτη ανταλλαγή απόψεων πάνω σε αυτό το φάκελο, ε, χαίρομαι το γεγονό ότι κάποια από τα θέματα τα οποία αναφερθήκαμε συμπεριλαμβάνονται συμπεριλαμβάνονται όπω ε, για παράδειγμα η προστασία των ευάλωτων ομάδων από την εκμετάλλευση, από την μετακίνηση σε ε, περιοχέ όπου υπάρχουν ε, διαμάχε, Έχουμε καταθέσει πάνω σε αυτά διάφορε τροπολογίε, όπω επίση και για την απασχόληση. Επίση, θέλουμε να δηλώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα δεν αντικαθιστά θέσει εργασία και γι' αυτό το λόγο ε, κατέθεσα δύο τροπολογίες ούτως ώστε όλες ε, οι ε, περιπτώσεις να είναι έμισθες και να πληρώνονται από τον οργανισμό που φιλοξενεί τους συμμετέχοντες Συνεχίζω επίσης να έχω τις αμφιβολίες μου όσον αφορά τη συμμετοχή του μη κερδοσκοπικού τομέα. Είναι σημαντικό επίσης ο κανονισμός να έχει ένα ξεκάθαρο ορισμό του εθελοντικού κομματιού, τους ώστε οι νέοι να έχουν πρόσβαση σε δυνατότητες εθελοντισμού που δεν θα χρησιμοποιηθούν ως αντικατάσταση ε, της πληρωμένης εργασίας για τους νέους. Ο εθελοντισμός δεν θα πρέπει να ε, αντικαθιστά την πληρωμένη εργασία, και, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει νέες δυνατότητες, νέες δεξιότητες και επίσης ε, είναι μια διαδικασία η οποία θα βοηθήσει ούτω ώστε να μεταφερθούν οι νέοι από, την, από τον εθελοντισμό στην ε, μελλοντική πληρωμένη εργασία και θα πρέπει να διασφαλιστεί επίσης η απασχόληση ε, και θα ήθελα να τονίσω ότι όλο αυτό θα πρέπει να γίνεται με ξεκάθαρους κανόνες και θα χαρώ να δω να τονιστεί το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη δεν θα αντικαθιστά και δεν θα αναμειχνύεται με άλλα προγράμματα εθελοντισμού και ενώ άλλα ε, προγράμματα όπω είναι το Erasmus Plus θα πρέπει να ενισχυθούν και ανησυχώ επίση όσον αφορά τη χρηματοδότηση που παίρνει χρήματα από άλλα προγράμματα τα οποία ήδη υπάρχουν και θα χαρώ να συνεργαστώ με την εισηγήτρια πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και... Η Τζιν Λάμπερτ ε, εκπροσωπεί του πράσινου, αλλά λείπει. Τον αντικαθιστά κάποιο. όχι. Τότε ο κ. Μαχτέ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό που είναι λυπηρό είναι ότι στην αρχή της δικής μου εισήγηση μιλήσατε στη θέση του εισηγητή και του ε, εκπροσώπου του SND. Αν σας είχα δώσει όμως δικό μου κείμενο για να με εκπροσωπήσετε, δεν είμαι βέβαιος ότι θα το διαβάζατε. Ε, για την εκπρόσωπο της Γκουε που είναι νέα, όπως και εγώ, θα ήθελα να σας πω ότι μια ιδρυτική ε, η συνθήκη της Ένωσης ορίζει την έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και ότι οι Βρυξέλλες είναι ένα παράρτημα. Το Στρασβούργο είναι η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και αν δεν σας αρέσει αν δεν σας αρέσει. Μπορεί κάθε φορά να το αφισβητείτε, αλλά είναι μέσα στις δυτικέ συνθήκες. Αλλά έχουμε τη συνήθεια με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση να διοργανώνουμε δημοψηφίσματα, τα οποία όταν είναι αρνητικά τα ξεχνάμε, τα ξεπερνούμε, τα ισοπεδώνουμε και περνάμε από τα κοινοβούλια. Τώρα, όσον αφορά αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ε, εκπρόσωπος της Άλτη που έφυγε δυστυχώς μας θύμισε πως έπρεπε να αποτελέσει για τους νέους μας μια πραγματική προστιθέμενη αξία κατά πρώτον και για τους πληθυσμούς που βοηθούνται θα έπρεπε να πρόκειται για μια πραγματική στήριξη και υπηρεσία κατά δεύτερο λόγο και διαπιστώνουμε ότι εμείς αμφιβάλλουμε πολύ για αυτή την προσθέμενη αξία και για την εξασφαλισμένη υποτιθέμενη πραγματική υπηρεσία. Εμείς θεωρούμε πως πρόκειται για ένα ακόμα μέσο να τονιστεί η κινητικότητα. Η κινητικότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε τα θεμέλια των εθνών που συναποτελούν αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι όλο ένα και περισσότερο άμορφα. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Αυτό που είναι το πιο σοβαρό είναι αυτό που, ε, που είπε και η πρόσωπος της ΓΟΕ. Πρόκειται για την υποαπασχόληση και τους ε, υπομισθούς. Κοιτάξτε το στόχο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης απευθύνεται στους νέους 18 με 30 ετών. 30 ετών νέοι 30 ετών. Μα μέχρι πότε είναι νέο κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 30, στα 35, στα 40. Είναι κρυπτοανεργία. Είμαστε νέοι από τα 18 μέχρι τα 25 και όπως είπε και η εκπρόσωπος της ΓΟΕ, έρασμος ναι, έρασμος συν για ολόκληρο τον κόσμο, όχι εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων που είναι άνεργοι και υποαμείβονται μέχρι τα 30 τους χρόνια είναι απαράδεκτη προτείνονται μία μάξιμουμ ε, ε, διάρκεια ενός έτους. Πάντως, η συμβολή της Κομισιόν δεν θα καλύψει παρά ένα έτος. Άρα, λοιπόν, δεν είναι ε, μόνιμες θέσεις, αλλά είναι υποβοηθούμενες θέσεις και υπάρχει ο κίνδυνος στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να μετατραπεί σε ένα εργαλείο απόκρυψης στοιχείων της ανεργίας των Ευρωπαίων νέων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, τι δίνουμε άρτων και θεάματα έτσι ώστε ο κόσμος να μην ξεγείρεται. Το αντίθετο ακριβώς από αυτό που συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία. Η αλληλεγγύη σας θυμίζω, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι πιο αποτελεσματική κοντά στην κοινότητα, ε, κοντά στην δική σου κοινότητα. Εάν κανείς εκτίθεται στους κινδύνους του ανθρωπιστικού τουρισμού, είναι πολύ επικίνδυνη όλη αυτή η διαδικασία. Και αυτό κάνετε, δημιουργείτε ε, μακρινά ταξίδια με αβέβαια αποτελέσματα και χωρίς να υπολογίσουμε και τις καταχρήσεις των ψευδομικίων που εκμεταλλεύονται γυναίκες και παιδιά. Και όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, με προπολογισμό 1,26 δις ευρώ. 1,26 δις ευρώ. Εσείς ακούτε τον κόσμο που γκρινιάζει, που παραπονιέται, λάβετε τον υπόψη και εγκαταλείψτε αμέσως αυτού του είδους ε, τα πολιτικά τεχνάσματα και δολώματα, αυτή την προπαγάνδα με κατεύθυνση τους νέους. Σας ευχαριστώ. Thank you, uh, Madam Lambert from the Greens. You arrived late, but it's your turn. Η κυρία Λάμπερτ από του Πράσινου, αν και καθυστερήσατε άλλα, δεν πειράζει, πάρτε το λόγο. Συγγνώμη ζητώ που καθυστέρησα, λέει η κυρία Λάμπερτ. Και νομίζω ότι πολλοί μόνο ε, κατανοούν ότι η σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας, η κατανόηση των άλλων χωρών, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ε, οι άνθρωποι στις άλλες χώρες είναι σημαντική. Και νομίζω ότι αυτό μαζί με το γεγονός ότι αυξάνονται ε, οι τάξεις εθνικισμού, λαϊκισμού και το καθεξής είναι κάτι που μας πρόχνει προς την κατεύθυνση αυτή. Οι τροπολογίες που καταθέσαμε σε ό,τι αφορά την έκθεση της κυρίας Κλούν που αποτελεί πάρα πολύ καλή βάση θεωρούμε έχουν να κάνουν ακριβώς με τα θέματα αυτά του να τονιστεί η φύση του εθροντισμού που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατανοούμε και εκτιμούμε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για τις δικλείδες ασφαλείας συνάδει αυτό και με τη δουλειά που έχουμε κάνει και σε άλλα σημεία εδώ στο Κοινοβούλιο. Και θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο έχει δυνατότητες να παρέχει προστιθέμενη αξία, αρκεί φυσικά ο προπολογισμό να είναι ειδικά για το πρόγραμμα αυτό, να μην αφαιρεθούν από αλλού αυτά κονδύλια αυτά. Προσβλέπουμε λοιπόν στη συνεργασία με την εισηγήτρια και να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα δώσει επιπρόσθετες ευκαιρίες για νέους που δεν έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές τέτοιες εμπειρίες που ασφαλώς και είναι πολύ σημαντικές για τα άτομα αυτά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Έχουμε εδώ και έναν εκπρόσωπο από τη Γενική Διεύθυνση τον κύριο Φραντ. Θέλετε να σχολιάσετε τα όσα ακούσατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τις προτινόμενες ε, τροπολογίες και τα σχόλια και να κάνω κάποιες ε, διευκρινήσεις για την πρόταση που υποβάλαμε. Θα θυμάστε ίσως ότι συνεργαστήκαμε για το τρέχον Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης σε ό,τι αφορά δηλαδή το έτος 2018-2020. Ο κανονισμός δημοσιεύθηκε μόλις τις αρχές του Οκτώβρη την επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δραστηριότητε και οι υπηρεσίες που αφαιρούνται από το Erasmus Plus και έχουν μπει στο σώμα αλληλεγγύης. Αυτό θα διτρηθεί και στο μέλλον. Άρα στο πρόγραμμα, όπως προτείνεται στο Erasmus Plus, δεν υπάρχουν εθελοντικές ε, δράσεις πλέον. Αυτές πλέον συμπεριλαμβάνονται στο, εθνικό, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η βάση τώρα της κατάρτισης της προτάσης μας ήταν ο συμβιβασμός που είχε πετύχει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Σώμα Τα στοιχεία που είχαμε καταφέρει να περάσουν για την πρόταση συμπεριλήφθησαν, αλλά προφανώς ε, η συμφωνία μετά από την σύναψη, από την δημοσίευση του κανονισμού και άρα υπάρχει κάποιο περιθώριο εκεί. Το θέμα τη ηλικία να το διευκρινίσω, γιατί συχνά μα ρωτάνε γιατί βάζουμε τα 30 έτη όριο. Γιατί. Να επιστήσω την προσοχή των αξιότιμων μέλων τη επιτροπή στα έγγραφα εργασία του 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι μέχρι την ηλικία των 30 ο κόσμος είναι ακόμα, έχει μόλις βγει από την, τον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ηλικία αυτή είναι 29-30 έτη ε, στο σημείο δηλαδή που ο κόσμο έχει τελειώσει, είναι, έχουν τελειώσει την εκπαίδευσή του, είναι 29-30 έτη. Άρα στο Erasmus Plus ως σημείο αναφορά, παραμένει αυτή η ηλικία 29-30 έτη. Όταν προτείναμε τον κανονισμό τώρα, ακολουθήσαμε λοιπόν την αρχή τη εναρμόνιση του κανονισμού στο βαθμό του δυνατού με, με τα άλλα προγράμματα χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό και αυτό Σχόλια εκτός μικροφώνου του, κυρία Μαρτά. Αυτό αποτυπώνεται και σε αλλαγέ στην πρόταση. Απαντάει η Επιτροπή. Δύο στοιχεία θα ήθελα να διευκρινίσω, πολύ σημαντικά. Συζητήθηκαν και με μεγάλο βαθμό λεπτομέρεια στην τρέχουσα διαπραγμάτευση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το θέμα τη υποκατάσταση θέσεων απασχόλησης. Η εθελοντικές ε, δραστηριότητες δεν μπορούν να οδηγήσουν σε υποκατάσταση πραγματικών θέσεων εργασία. Υπάρχουν διάφορε δικλείδε ε, ασφαλεία. Και επαναλαμβάνω την αρχή ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει αντικατάσταση ε, θέσεων απασχόληση ή να καταλήξουμε σε δουλειέ χωρί πληρωμή. Δεύτερο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι η πτυχή της συμπερίληψης και πολλοί συνάδελφοι. Και εδώ και σε άλλες επιτροπές επιμένουν ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι ανοιχτό. Ανοιχτό σε συμμετοχή σε διάφορες ε, ομάδες νέους Ευρωπαίους δηλαδή. Να μην εξαιρείται κανείς. Υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική συμπερίληψης Έχουμε συγκεκριμένο μορφότυπο και χρηματοδότηση για τη συμμετοχή όσο πιο πολλών νερών Ευρωπαίων γίνεται. Τέλος, διάφορες ομάδες ζητήσαν να υπάρχει μια διαδικασία για ποιοτική σφραγίδα σε ό,τι αφορά εθελοντικές θέσεις απασχόλησης και πρακτικές. Εμεί θέλαμε μία τέτοια σφραγίδα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων μορφοτύπων. Και γιατί το λέω αυτό. Μπορεί να φαίνεται ότι μία οργάνωση θέλει να πάρει την σφραγίδα ποιότητα και για εθελοντισμό και για μία πρακτική και αυτό θα πρέπει να μπορεί να το πετύχει και μάλιστα με έναν ενιαίο τρόπο. Άρα, συνοψίζοντας, ευχαριστώ και πάλι για την πρόταση και ελπίζω ότι μαζί θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ τον κανονισμό μας. Thank you. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι έχουμε κάποιον και από την Επιτροπή. Όχι. να συστηθώ Ρόμπερτ ε, Φράντσαϊν και εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Γενική Διεύθυνση Απασχο... Ε, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Ωραία λέει η Πρόεδρος. Συγγνώμη που η κυρία Κλούνε δεν μπορούσε να παρευρεθεί, ίσως ε, ε, να μπορέσουμε να ξεκλέψουμε κάποια λεπτά την, στην επόμενη συνάντησή μας, ούτως ώστε να μπορέσει και η ίδια να συνεισφέρει ε, στην ενημέρωση και στη συζήτηση, διότι αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία εισάγαμε, εφεύραμε θα μπορούσαμε να πούμε και για το οποίο έχουμε εργαστεί ιδιαιτέρως ε, στην Επιτροπή μας. Θα το τονίσουμε λοιπόν ε, θα το σημειώσουμε ούτως ώστε η κυρία Κλούνε στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Απασχόλησης ε, να μπορέσει να ε, παρευρεθεί και να συζητήσει και αυτό το θέμα. Η υιοθέτηση στην ΕΜΠΛ είναι για τις 3 Δεκεμβρίου ενώ στην Επιτροπή Κούλτ για τις 4 Φεβρουαρίου και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που αφορά το Εράσμους, το ε, πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πάβελ. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, που, δίνετε, που δείξατε ενδιαφέρον για το φάκελο Εράσμους. Έχουμε συνολικά 303 τροπολογίες ε, και τώρα θα εργαστούμε πάνω σε αυτές ώστε να βελτιώσουμε την ε, πρόταση. Το ημερολόγιο μας έχει αναθεωρηθεί. Η ψηφοφορία θα γίνει τώρα στις 3 Δεκεμβρίου το ημερολόγιο της Κάλτσατ άλλαξε όμως και μάλλον θα γίνει στις 20-21 ε, Ιανουαρίου. Ευχαριστώ τους Κιώδης ε, που αποδέχθηκαν τις αλλαγές ε, στις ημερομηνίες για την Επιτροπή ΕΜΠΛ. Με βάση τις αλλαγές στην Επιτροπή ΚΑΛΤ είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την πρώτη μας συνάντηση στο Στρασβούργο και ανυπομονώ να ακολουθήσουν και οι επόμενες. Και τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, σχόλιο εκτός μικροφώνου, είχαμε συνάντηση απαντά στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ αρνούμαι να πάω. Ε, για λόγους αρχής. We take notice Σημειώνουμε τα σχόλιά σας. Οι προτεραιότητες που έχουμε τώρα όσον αφορά το κομμάτι της απασχόλησης ε, είναι η καλύτερη προώθηση ε, του προγράμματος ε, στην επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων, το οποίο θα πρέπει να φαίνεται στην κατανομή του προπολογισμού όσον αφορά και, την, και το πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρχει ευέλικτη χρηματοδότηση, ούτως ώστε να επιτύχουμε αυτή τη σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα Erasmus+. Θα πρέπει επίση να προωθήσουμε ε, την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων και να προωθήσουμε επίση την ευελιξία. Επίση, ο περιεκτικό χαρακτήρα του προγράμματο ε, προσφέρει την ε, ε, προσέγγιση σε ανθρώπους ε, με λιγότερες δυνατότητες, το οποίο επίσης μας απασχολεί. Η υποστήριξη ανθρώπων με λιγότερες δυνατότητες θα πρέπει να είναι τόσο ε, διαρθρωτική όσο και οικονομική. Επίση, για να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα είναι δίκαιο και προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερου Ευρωπαίου, ε, τα επίπεδα οικονομική ε, υποστήριξη, όπω είναι για παράδειγμα ε, καταποκοπή ποσά, υποτροφίε, θα πρέπει να εξετάζονται συνεχώ και να προσαρμόζονται ούτω ώστε να υποστηρίζουν τα έξοδα διαβίωση τη χώρα φιλοξενία. Τέταρτον, για να διασφαλίσουμε ε, την θετική επιρροή στους Ευρωπαίους πολίτες θα πρέπει να ζητήσουμε το πρόγραμμα να διασφαλίσει κινητικότητα με βάση τις αρχές ε, της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Χάρτας Κινητικότητας ε, και θα πρέπει να υποστηρίζει την μετακίνηση καθώς επίσης και ένα ξεκάθαρο σχέδιο μάθησης. Κάθε πλαίσιο μάθησης θα πρέπει να αξιολογείται και να αναγνωρίζεται και γι' αυτό το λόγο ζητούμε την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτελεσματικής και ποιοτικής ε, μαθητείας ε, καθώς επίσης και κάθε άλλο ευρωπαϊκό εργαλείο το οποίο συνεισφέρει στην μάθηση στο εξωτερικό και την αξιολόγηση ε, των, ε, της μάθησης. Πιστεύουμε ότι με όλα αυτά μπορούμε να συνεισφέρουμε στη βελτίωση του προγράμματος Erasmus Plus και κατά συνέπεια να υποστηρίξουμε την προσωπική και επαγγελματική ανέλυξη των πολιτών μας. Ανυπομονώ λοιπόν να εργαστώ μαζί σας πάνω σε αυτό το φάκελο. Αύριο έχουμε μια συνάντηση σκιωδών και την Τετάρτη επίσης άλλη μια συνάντηση και αν ε, τα καταφέρουμε ως τότε, τότε πιστεύω ότι η ψηφοφορία σίγουρα θα μπορέσει να γίνει την 3η Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Pavel. Ε, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πάβελ. Ο κύριος Μαν από το ΕΛΚ είναι καθοδόν. Όσο τον περιμένουμε θα ακούσουμε την κυρία Στίβενς από το ECR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και την πολύ επικοδομητική στάση. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερω ε, το πρόγραμμα Erasmus Plus και χαίρομαι ιδιαίτερω που ο εισηγητή ε, θέλει να ενισχύσει το πρόγραμμα αυτά χωρί ε, περίτε επιβαρύνσεις. Όποιος έχει ωφεληθεί από την εμπειρία του Εράσμους έχει πραγματικά πολλά να πει. Δίνει πολλές ευκαιρίες και προσωπικής ανάπτυξης και στην επαγγελματική ανάπτυξη και είναι πιο εύκολο να βρει δουλειά στο μέλλον. Χαιρόμαστε λοιπόν που το Erasmus είναι προσβάσιμο για όλους τους νέους μεταξύ των οποίων και τους νέους με αναπηρία. Αυτό ωφελεί όχι μόνο τα άτομα, αλλά και τις κοινωνίες στο σύνολό της. Όσο δημοφιλές όμως και αν είναι το πρόγραμμα Εράσμου, στο παρελθόν φάση αποτελεί, μάλλον οι νέοι με αναπηρία που το χρησιμοποιούν είναι κάτω από 1% και εγώ προσωπικά το είδα ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα προσβασιμότητας έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσει ένα νέο ε, κοφάλαλο ε, το πρόγραμμα Εράσμου, γιατί θα πρέπει να πληρώσει τα έξοδα του διερμηνέα, του νοητική. Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφωθεί το πρόγραμμα με ε, συμπεριληπτικό τρόπο και αυτό δεν μπορεί να είναι και ένα λόγια μόνο και διαπιστώνω με χαρά ότι ο εισηγητή κάνει ό,τι μπορεί για να μεταφραστούν όλα αυτά σε συγκεκριμένε δράσει και θα ήθελα να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα άτομα με αναπηρία. Ούτε τα έξοδα συμπερίληψη ε, σημαίνει ότι μπορεί να απορρίπτουν τέτοιε αιτήσει. Θα πρέπει να ορίσουμε τι χρηματοδοτικές ε, απαιτήσει και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πραγματικά επιτυχάνεται αυτή η συμπερίληψη. Προτείνω λοιπόν να γίνεται σαφής αναφορά δικτών ε, αποτελεσματικότητας για νέους από λιγότερο εύπορες ε, ομάδες. Και τέλος να εκφράσω και μια ανησυχία. Η παιδεία αποτελεί κατά πρώτο λόγο αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό έχουν συμφωνήσει και βρήσει σε συνθήκες στα κράτη-μέλη και με ιδιαίτερη προσεκτική σε ό,τι αφορά την ιδέα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Δεν ε, σημαίνει αυτό φυσικά ότι δεν υποστηρίζω την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το εράσμος δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται τόσο πολύ στο πόσοι συμμετέχουν, αλλά στην ποιότητα και θα ήθελα να τονίσω και την ε, Discover EU πρωτοβουλία. Εδώ το υπογραμμίζω το θέμα αυτό. Και υποστηρίζω τον εισηγητή στην ε, αξίωσή του για αύξηση των κονδυλίων και επίσης ε, να πούμε ότι η χρηματοδότηση πάντα θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένε ανάγκε και σε αύξηση τη αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Προσβλέπω στην συνεργασία με τον εισηγητή και με του υπόλοιπου κοιόδες για να γίνει ένα καλό βήμα προ ένα πιο συμπεριληπτικό και πιο σωστό πρόγραμμα Εράσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Στίβεντ. Ακούσαμε τον εισηγητή, την κυρία Στίβενς και τώρα κύριε Μαν η σειρά σας παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Παρατηρώ ότι όταν συγκρίνουμε ε, την 17η ε, δεκάτου ε, και την πρώτη συζήτηση τότε, οι ελπίδες ήταν μεγάλες τότε και όντως ε, εκπληρώθηκαν οι ελπίδες μας. Αυτό είναι ένα γενικό ε, σχόλιο. Το εράσμος δεν θα πρέπει να αφορά μονάχα το πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα και τους ε, συμμετέχοντες στην ε, προγράμματα επαγγελματικής ε, κατάρτισης και γι' αυτό το λόγο έχουμε διάφορες τροπολογίες, ούτως ώστε στις διαπραγματεύσεις την Τετάρτη να έχουμε δυνατότητες συμβιβασμού. Έχω κάποια σημεία όμως, τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε. Αρχικά όσον αφορά το θέμα, το άρθρο 2 παράγραφο 1 Εκεί αναφέρεται ότι ο βασικός στόχος της ε, εκπαίδευσης ανηλίκων είναι η κοινωνική συμπερίληψη ε, και ίσως θα έπρεπε να αναφερθούμε εκεί στο social market ε, και όχι μονάχα στο labor market. Και το άλλο θέμα, ο συνάδελφος Μπέκερ έκανε μια, ε, τρο, μια τροπολογία όπου θα ήθελε ε, να ε, αναφέρεται και η ηλικία, η τροπολογία 159 νομίζω, δεν μπόρεσα να τη βρω όμως, αν μπορούμε να τη βρούμε δεν είναι τόσο σημαντικό βέβαια. Στο άρθρο 2 παράγραφο 1 έχουμε την συνεργασία μεταξύ των τομέα. Cross-sector cooperation είναι μια έννοια που δεν χρησιμοποιήθηκε πριν, όπως επίσης και οι λέξεις ε, mobility providers, πάροχος κινητικότητας. Θα μπορούσατε λοιπόν να αιτιολογήσετε για ποιο λόγο ξαφνικά χρησιμοποιούνται αυτοί οι δύο όροι ε, τη στιγμή που στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Τρίτον, ε, έκανα ε, μία ανθρωπολογία 205 θα ήθελα ένα άρθρο όπου υποστηρίζουμε την δημοκρατική κατανόηση. Αυτή τη στιγμή λέμε για συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο. Μήπως αυτό είναι λίγο. Ε, όταν μιλάμε για δημοκρατία, τη δυνατότητα οι νέοι να λένε πως είναι οι δομές καταρτισμένες σε μια δημοκρατία. Ε, για ποιο λόγο υπάρχουν και η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι έρχονται και προστίθενται. Ε, η κατανόηση της δημοκρατία σημαίνει κάτι περισσότερο. Να λέμε για ποιο λόγο είναι κάτι τόσο πολύτιμο η δημοκρατία. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι μονάχα το participation in democratic life, συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή, είναι κάτι πολύ λίγο. Επίσης θα μπορέσουμε να έχουμε ε, κάποιες δραστηριότητες για παράδειγμα. Οπότε λοιπόν θα ήθελα να συμπεριληφθεί αυτό στην ε, συμβιβαστική. και επίσης υπήρξαν κάποιες ε, προτάσεις που θα θέλαμε να συμπεριληφθούν από τη συνάδελφο Αγνιέσκα Βοσλοφσκάια ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, και οι ε, ηλικιωμένοι μαθητευόμενοι, αυτοί οι οποίοι ε, σπουδάζουν, μαθαίνουν σε μεγαλύτερη ηλικία ε, θα, υπάρχει μια τροπολογία για αυτό, όμως ε, αυτό ακριβώς το κομμάτι δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε μια αιτιολογική σκέψη πάνω σε αυτό. Αυτά λοιπόν κατά βάση είναι οι βασικότερες σκέψεις που έχω. Ε, ένα τελευταίο στην τροπολογία 10 έχουμε το θέμα ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Όμως το Εράσμος δεν υπάρχει για να συζητήσουμε το θέμα του μισθού ε, αφορά την, ε, το ζήτημα του κόστους ε, για παράδειγμα αλλά δεν νομίζω ότι το equal pay for equal work έχει θέση εδώ. ξέρω ότι διαφορετική η κατάσταση στη Ρουμανία και διαφορετική στη Βιλανδία και θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη ε, κατανομή των χρημάτων όμως δεν νομίζω ότι αυτός ο όρος ταιριάζει εδώ πέρα. Ή ε, θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ καλή ε, εργασία. Δύο τροπολογίες δεν τις κατάλαβε ε, γιατί ήταν στα ουγγρικά. Βέβαια, εσύ σίγουρα θα μπορούσες να τις καταλάβεις καλύτερα. Συνολικά, λοιπόν, πιστεύω ότι όσον αφορά ε, την Επιτροπή μας πηγαίνουμε πολύ καλά. Ευελπιστώ το ίδιο να κάνει και η Επιτροπή Πολιτισμού πάνω σε αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάν. Δεν υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της αλτε ούτε της Γκουε NGL. Πράσινη, όχι. Δεν προσωπείται το κύριο Μέτερνιχτ σήμερα. Η FDA η D κανέναν και ούτε το INF. Το σημαίνει ότι θα δώσω το λόγο στον κύριο Πάβελ. Στα γερμανικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια που μας είπατε. Και σε ό,τι αφορά τις ασάφειες, είχα μία συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητήσαμε τα θέματα του ορισμών, τα οποία τα αναφέρατε και εσείς. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι αποσύρθηκαν. Αλλά θα το κάνουμε αύριο στις πρώτες συζητήσεις μας και την Τετάρτη θα οργανωθεί η δεύτερη συνάντηση σε ό,τι αφορά τα θέματα δημοκρατίας. Ε, το τονίσαμε αυτό και στις τελογικές σκέψεις. Σε ό,τι αφορά τον ε, διαστομένο διάλογο των νέων, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και ενδεχομένω να βρούμε και περαιτέρω λύσεις αν σας αρκεί αυτό που έχουμε γράψει. Νομίζω ότι δεν απέχουν πολύ οι απόψεις μας και είμαι αισιόδοξο ότι και αύριο και μεθαύριο θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το μεγαλύτερο τμήμα των αποφάσεων που έχουμε να λάβουμε. Μην σας πω και όλες και πιστεύω ότι μας ε, περιμένει εύκολη και παραγωγική και ομαλή ε, συνεργασία. Τα σημείωσα όλα με τους συναδέλφους και θα σας κάνουμε τις προτάσεις μας αύριο. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, the will be... Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αποσχόλησης θα γίνει στις 3 ε, Δεκεμβρίου, ενώ στην Κούλτ στις 22 Ιανουαρίου. Αυτά για απόψε. Έχουμε αύριο τρεις ώρες ψηφοφορίας. Οπότε ήταν καλό που είχαμε ένα σύντομο ζέσταμα σήμερα. Θα χρειαστούμε όλη μας την ενέργεια για να ε, συγκεντρωθούμε αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ λήξη της συνεδρίασης. I <laughs>